ερχόμαστε στις επεξηγήσεις ψήφου και αρχίζουμε από το ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουκρανία και την κατάσταση ε, και τις εξελίξεις της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Η κυρία Τζουφρίντα είναι πρώτη στις επεξηγήσεις ψήφου. Για ένα λεπτό παρακαλώ, σας θυμίζω. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα διότι πρέπει να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια για να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας χωρίς να λησμονούμε ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια διπλωματική λύση και πολιτική λύση που όλοι ευχόμεθα ότι θα εξευρεθεί τάχιστα θα πρέπει τάχιστα να βρεθεί μια ειρηνική διέξοδο, ταυτόχρονα να αφήσουμε ανοιχτέ διάβλου επικοινωνίε και να είμαστε έτοιμοι να επανεξετάσουμε σε περίπτωση θετική τροφοδότηση, κυρώσει και τι συνέπειε έχουν. Λαμβάνοντα υπόψη συμβαίνει στη Γεωργία, στη χώρα μου, κυρία Τζουφρίντα διακόπτη πρόεδρο. Πηγαίνετε πιο αργά για να μπορούν να σα προλαβαίνουν οι διερμηνεί και έχοντας ακούσει την αποφασιστικότητα της, ε, του Επιτρόπου Τσόλος επιμένω παρόλα αυτά στην ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι να είναι σαφείς διότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να ευεργητηθεί από ενισχύσεις σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες παραγωγικές που έχει και μπροστά στα μάτια όλων βλέπουμε ότι οι πόροι είναι ανεπαρκείς και χρειάζονται μεγαλύτερα κονδύλια και για αυτό το σκοπό για να φέρω παράδειγμα την Ιταλία, να επενθυμίσω ότι οι ζημιέ μας φτάνουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ από τις κυρώσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρντίνη, επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να εξηγήσω γιατί εμείς δυστυχώς δεν μπορέσαμε να υπερψηφίσουμε αλλά έχουμε απόσχη από αυτή τη σημαντική, ε, σημαντικό ψήφισμα. Από τη μία πλευρά βέβαια συμμεριζόμαστε τις τεράστιες ανησυχίες για το γειτονικό μας ουκρανικό λαό, για τις δραματικές στιγμές που ζει και συμμεριζόμαστε όλο το τμήμα αυτό που αφορά την υποστήριξη και την εξέβρεση λύσης και το ότι πρέπει να καλυφθούν και οι τομεί Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πληγεί οικονομική. Υπάρχουν και άλλα σημεία πολύ σημαντικά όμω που δεν μπορούμε να συμμεριστούμε, όπω το σημείο που αφορά τον ενεργειακό τομέα, όπου μιλάμε για ακύρωση των συμφωνιών με τη Ρωσία όπως και το σχέδιο στο πρόγραμμα South Stream. Και γι' αυτό με θρύψη μας έχουμε απόσχεια, αλλά επίσης με διπλωματική ε, οδός να οδηγήσει σε μια λύση, σε μια πολιτική λύση που αυτή πρέπει να είναι, μια πολιτική λύση. Ευχαριστώ κυρία Καρδίνη. Η κυρία Ζντανόκα είναι επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα. Είμαι βέβαια ότι σειρά συναδέλφων εξακολουθούν κάθε φορά να βγάζουν τέτοια κείμενα που βασίζονται σε μονομερείς ε, προσεγγίσεις. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, σε πολλές εκθέσεις διεθνών ΜΚΟ και της Διεθνούς Αμνηστίας ιδιαίτερα, η Ουκρανική κυβέρνηση κατηγορείται ε, ότι παραβιάζει σκληρά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, με λεγόμενες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Το αρχικό κείμενο, παράγραφος 2 του κείμενου μας, του ψηφίσματος αναφέρεται μεν σε αυτή την έκθεση αλλά μιλά για παραβιάσεις που γίνονται κυρίως ε, από ε, αποσχιστές και το τακτικό ρωσικό στρατό ε, και κάποια φορά μπορεί να είναι και κανένας Ουκρανός. Είναι πολύ στρεβλή αυτή η εικόνα που δίνεται από τα ευρήματα των ΜΚΟ και αποδυναμώθηκε από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου η πραγματική εικόνα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πιετικά Mrs. είναι. Κυρία είναι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Ε, είναι γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσαμε ε, για μια κοινή γραμμή απέναντι στην περιφέρεια αυτή και σε σχέση με τη δική μας ασφάλεια. Πρέπει να έχουμε μια συνεκτική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, σύραξη. Επίσης θα πρέπει να ενισχύουμε και την οικονομική μας πολιτική στην περιφέρεια αυτή πάντα. Άρα θα πρέπει η κατάσταση να σταθεροποιηθεί και εμείς να σταθεροποιήσουμε τις σχέσεις μας και να τις εξομαλύνουμε και με τη Ρωσία. Αυτή η Ουκρανική κρίση είναι για την πολιτική ασφαλείας ε, ότι και η χρηματοοικονομική κρίση για την οικονομική μας πολιτική. Και τώρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε μία ενιαία γραμμή και μία ενιαία φωνή. Οι κυρώσεις είναι ένα μικρό βήμα πρόοδου, είναι καλές, ας ελπίσουμε όμως να αποδώσουν κιόλας. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στο επόμενο ψήφισμα. Αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση στην έξαρση τη επιδημία έμπολα. Η κυρία Ζαμπόσκα είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα πολύ σαφέ ε, και ξεκάθαρο ψήφισμα ε, απέναντι σε αυτή την ε, τόσο σοβαρή ασθένεια. Είχαμε αυτό το κρούσμα έμπολα, είναι πάρα πολύ περίπλοκη η κατάσταση και οι συνέπειες ανυπολόγιστες. Σιγά σιγά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση. Δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Δυτικής Αφρικής, είναι παγκόσμιο πλέον το πρόβλημα. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε τα εξής δύο πράγματα. Ε, από κοινού να αναπτύξουμε μέσα αντιμετώπισης και φάρμακα και δεύτερον η καραντίνα και τα διάφορα υγειονομικά μέτρα να ε, γίνονται να εφαρμόζονται σωστά. Μόνο έτσι θα έχουμε πραγματική υγεία και ε, ο κόσμος θα πρέπει να εμπιστεύεται το υγειονομικό προσωπικό και την κυβέρνηση. Δυστυχώς ε, στη Λιβερία αυτό δεν συμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να σταθεροποιηθεί και η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι κίνδυνοι για την υγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να φοβίζουμε τον κόσμο. Ξέρουμε ότι σε παγκοσμιοποιημένο κόσμο οι άνθρωποι και τα αγαθά κινούνται ελεύθερα. Εξίσου και κίνδυνοι για την υγεία. Είναι πλέον παγκόσμια μορφή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώ, θα πρέπει να είναι πιο ταχεία στην αντίδρασή της σε περίπτωση παγκοσμίων τέτοιων κινδύνων για την υγεία και κινδύνων για επιμόλυνση. Όσον αφορά την έμπολα, Φαίνεται ότι τα ληφθέντα μέτρα αρκούν. Βλέποντας πόσο επικίνδυνη είναι η ασθένεια, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει σύστημα ταχείας αντίδρασης για περίπτωση όλων των μολυσματικών ασθενειών. Από τη στιγμή που είναι επικίνδυνε αυτέ οι ασθένειε. Ευχαριστώ. Πάμε στην επεξήγηση ψήφων για την κατάσταση του Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση τη ISIS. πρώτο ομιλητής, η κυρία Αρνούτου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που επιτέλους ενδιαφερόμαστε για τη μοίρα των μειονοτήτων και κυρίως των χριστιανών στον εγγύς Ανατολή. Αλλά είναι πολύ καθυστερημένη δυστυχώς αυτή η προσέγγιση και επιδεινώνεται από την, από την επίθεση των Αμερικανών στο Ιράκ εδώ και χρόνια. Λοιπόν, η, οι αντάρτες του ISIS είναι πάρα πολύ βίαιοι και ε, βλάπτουν τους πάντες. Πώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πολεμούμε ε, τους μεν υποστηρίζοντας τελικά τις λάθος δυνάμεις. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα μπορούν να ανέχονται η Τουρκία ε, να, ενισχύει τελικά και να εκπαιδεύει και να εξοπλίζει τα μέλη της ISIS και να δέχεται το πετρέλαιο που πολλούν και να διοργανώνεται η στρατολόγηση στο δρόμο. Πέρα από τις συνηθισμένες χειρονομίες που κάνουμε θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν τα σαφερές θέσεις κατά όλων των Ισλαμιστών σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Συρίας και του Ιράκ. Στη συνέχεια η κυρία Ντότς, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί από τις οργανικές δολοφονίες που είδαμε πρόσφατα στην Μέση Ανατολή και οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας πάνε στους, ε, στις οικογένειες εκείνων που έχουν πληγεί και με την οικογένεια του Άλαν Χένιγκεν και τον ίδιο τον Άλαν Χένιγκ που αντιμετωπίζει ε, φοβερή απειλή τις τελευταίες μέρες. Δεν πρόκειται μόνο περί αυτού, αλλά δολοφονούνται χριστιανικές κοινότητες στη Συρία και στο Ιράκ. Είναι επιτακτικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει μέσα αποτελεσματικά για να προστατεύσει τους χριστιανούς, σε ενικές μειονότητες σε όλη τη Μέση Ανατολή. Επίσης, θα... οι σκέψεις μου στρέφονται επίσης προς την πρόσφατα αποδημία του Λόρδου Μπανσάιντ, που εκπροσωπούσε την εκλογική μου περιφέρεια στο Κοινοβούλιο ανάμεσα στο 1979 και το 2004. Ήταν μεγάλος πρέσβης της χριστιανοσύνης, καθώς και υπέρθερμος υπερασπιστής της Βόρειας Ιρλανδίας. Η δουλειά του εδώ οδήγησε σε ευρωπαϊκή υποστήριξη για χρηματοδότηση ε, για την ειρήνη στην εκλογική περιφέρεια. Εμείς δεν θα δούμε κάποιον παρόμοιο στην Βόρεια Ιρλανδία ούτε στην Ευρώπη. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας πάνε στην σύζυγό του και στην οικογένειά του. Ευχαριστώ. Επόμενος, η κυρία Πιτήρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπερψήφισα και βέβαια υπέγραψε και το ψήφισμα αυτό, διότι βλέπουν τους τελευταίους μήνες πολύ σοπαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αιματοχυσία. Ε, ε, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, βλέπουμε τη δίωξη των αμάχων, ε, κυρίως δε των χριστιανών. Είναι πάρα πολύ η κατάσταση. Έχουμε 1,2 εκατομμύρια εκτοπιστέντες και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που χρειάζονται επιγόντως ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε συνεχώς ε, εξισλαμισμούς. Ε, το έχει πει και ο Πατριάρχης ότι ε, είναι κάτι για το οποίο όλοι οι μουσουλμάνοι θα έπρεπε να τρέπονται αυτά που βλέπουμε δηλαδή στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό θα πρέπει αυτού του είδους τις δολοφονίες να τις σταματήσουμε. Το συντομότερο δυνατό ελεύθερο η ελευθερία έκφρασης λόγου, πεπιθήσεων είναι ε, κάτι που θα έπρεπε να είναι γενές δικαίωμα κάθε ανθρώπινου πλάσματος. Δεν μπορούμε να στερεί κανείς αυτό το δικαίωμα, ε, γιατί τέλος είναι καταδικασμένος. Ευχαριστώ. Επόμενο μιλητή λεπρό ο κύριο Ζόγκορ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση τώρα και τη Συρία δημιουργεί πολύ σημαντικέ γεωστρατηγικέ ε, και πολιτικέ προκλήσει Βλέπουμε επίσης και μια τρομερή ανθρωπιστική κρίση για ευάλωτες ομάδες όπως θρησκευτικέ εθνικές μειονότητες, γυναίκες, παιδιά που δυσανάλογα πλήττονται από τις βαρβαρότητες του Ισλαμικού κράτους. Χρειάζεται γρήγορη, συντονισμένη δράση από τη διεθνή κοινότητα. Είναι σημαντικό για θρησκευτικού λόγους στη Μέση Ανατολή να καταδικαστεί η δράση του Ισλαμικού κράτους ε, με τον πλέον απερίφραστο τρόπο. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των ομάδων στο Ιράκ και ελπίζω η νέα κυβέρνηση Αλμπάντη να είναι και να βγει προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι η Ιρακινή κυβέρνηση θα πρέπει να επανεισαγάγει την έννοια ε, της ε, αλληλέγγυας ή μάλλον της ε, ηθαγένειας προς όλους, ε, ώστε όλοι οι πολίτες στη χώρα είναι ίσοι. Ευχαριστώ πολύ τελευταία ομιλητή για το θέμα αυτό, η πρόεδρος είναι η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Η πρόταση ψηφίσματος για την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία δεν αναφέρει σχεδόν καθόλου τους χριστιανούς. Αυτή όμως είναι ε, ο βασικός στόχος ε, ε, των βίαιων διώξεων αυτών των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους. Καταφέραμε στο κοινό ψήφισμα βέβαια να συμπεριλάβουμε δύο παραγράφους που αναφέρονται στη χριστιανική μειονότητα για την περιοχή αυτή και συγχαίρω τους διαπραγματευτές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και για την προσέγγιση που υιοθέτησαν. Ευτυχώ το κοινοβούλιο τελικά κατάφερε να εκφράσει την αλληλεγγύη του προ τι χριστιανικέ αυτέ κοινότητε που στι χώρε, στι πατρίδε του απειλούνται, διώκονται, απειλούνται με εκρίζωση. Λόγω της ε, θρησκείας τους, λόγω των πιστεύω τους, διώκονται, τους στερούνται τα βασικά δικαιώματα αναγκάζονται να γίνουν πρόσφυγες. Χαίρομαι πολύ που καταφέραμε να τονίσουμε την οδύνη τους, τα βάσανά τους και αυτό το ψήφισμα είναι το πρώτο βήμα για να επανέλθουν οι πρόσφυγες ε, αυτοί οι χριστιανοί στις χώρες τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο ψήφισμα. Κατάσταση στη Λιβύη. Ε, Ένα ομιλητή, μόνο ο κύριο Σαφχάουζε, έχει ζητήσει να κάνει επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η ομάδα μου και εγώ υπερψηφίσαμε το ψήφισμα αυτό γιατί λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στην καταστροφική κατάσταση στη Λιβύη και υπογραμμίζει και τα προβλήματα που γνωρίζουμε αλλά θα έπρεπε και να τα πούμε για την κυκλοφορία των όπλων, την παρουσία τρομοκρατικών ομάδων και μαζική μετανάστευση προς τις Ιταλικές ακτές. Ωστόσο θα θέλαμε να υπογραμμιστεί εδώ και ο ρόλος της Γαλλίας που είναι δυστυχώς η χώρα μου αλλά και του ΝΑΤΟ που βήθησε τη Λιβύη σε αυτή την κόλαση. Και εμείς θα θέλαμε να υπογραμμιστεί επίσης ότι η Λιβύη πάνω απ' όλα είναι θύμα αυτής της τυχοδιοκτικής διπλωματίας, για να μην πω τίποτα άλλο, της Ευρώπης και της Δύσης. Και αυτή τη στιγμή είναι αδιέξοδη κατάσταση και δεν υπάρχει βιώσιμη λύση. Και τώρα ε, προχωρούμε στην επεξήγηση ψήφου για το ψήφισμα σχετικά με τη Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Ο κύριος Κάρτη πρώτος. Εγώ καταψήφισα το κοινό ψήφισμα για την Παλαιστίνη διότι πιστεύω ότι στέλνει ένα μήνυμα ιδιαίτερα προς το Ισραήλ ότι μπορεί να συνεχίσει να κάνει τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων ε, ε, ατιμόρυτο. Οι λαοί της Ευρώπης θα απογοητευθούν μαθαίνοντας ότι ε, πολλοί Ιρλανδοί ε, στο Κοινοβούλιο ψήφισαν αυτό το ψήφισμα και καταψήφισαν την απελευθέρωση ε, εκλεγμένων ε, Παλαιστινίων που κρατούνται άδικα. Ε, επίσης, να διερευνηθούν τα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της τελευταίας Ισραηλινής επίθεσης. Το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης μιλάει για πάγωμα της Συμφωνίας όσο συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ και θα ζητούσαμε αποζημίωση από το Ισραήλ για προγράμματα και έργα που έχει έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ πρόσφατα κατέστρεψε με την επίθεση στη Γάζα το Ισραήλ. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ε, ε φέτος που είναι και επέτειος ε, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ε, ένα σύμβολο ειρήνης ενώ ένα σύμβολο αδράνειας απέναντι σε ένα παράνομο πόλεμο και την επίθεση κατά του Παλαιστινιακού λαού. Ευχαριστώ η κυρία Ντότς. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχουμε πολλές πτυχές που αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα των, της απάντησης που δίνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή αυτή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υποστηρίξουμε το κυριαρχικό δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τα σύνορά του και το λαό του από την τρομοκρατία. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη τα τεράστια δεινά που περνά ο λαός της Γάζας, που είναι άμεσο αποτέλεσμα της επιχείρησης και θα πρέπει να δράσουμε και να βοηθήσουμε. Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που είχε επιχείρηση στην ασφάλεια των Ισραηλικών των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε περίπου 240 καταγγελίες επεισοδίων αντισημιτικών τον Ιούλιο, όσο κλιμακωνόταν οι μάχες. Αυτού του είδους αδικημάτων και εγκλημάτων μίσους είναι απαράδεκτα σαν Ευρωβουλευτές και σαν Κοινοβούλιο. Είναι ζωτικό, ζωτική σημασία να στέλνουμε ένα μήνυμα στην Ευρώπη, δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ε, θρησκευτική ανοχή, η ανεξιθρησκεία. Ο κ. Σουρτασούν είναι επόμενο ομιλητή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα αυτό το οποίο συμβαίνει και έχει ήδη συμβεί στη Γάζα. Αντιμετωπίζουμε πραγματικά εγκλήματα κρατικά που γίνονται σε αυτή τη ε, φυλακή, τη Γάζα δηλαδή. Ε, σφαγιάζει το πληθυσμό τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί αυτή ε, την... δεν μπορεί να συνεχιστεί μάλλον να έχει ε, τηρεί πολιτική των αποστάσεων. Δεν είναι δυνατόν να τηρείται μια τέτοια πολιτική. Έξω και εμεί ψηφίσαμε κατά αυτού του ψηφίσματο που τη συνεχίζει. Θέλουμε να πάψει πραγματικά ο αποκλεισμό και η κατοχή. Δεύτερον, ε, να πάψουν οι παράνομοι επικισμοί και η παράνομη κατοχή αυτών των εδαφών που πλήττει του αγρότε. Τρίτον, να φτάσει και να, εφαρμοστεί, και να δοθεί εκεί που πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια για το Παλαιστινικό Συμβούλιο ε, και τους κρατούμενους να απελευθερωθούν. Επίσης, η Εθνής κοινότητα πρέπει να ε, ερευνήσει ε, για εγκλήματα πολέμου τους ηγέτες του Ισραήλ. Θα πρέπει τη Συμφωνία Σύνδεσης, το άρθρο 2, να δούμε αν μπορούμε να αναστείλουμε τη βοήθεια και την χρηματοδότηση σχεδίων που φέρνει σε πέρα στο Ισραήλ. Θα πρέπει, επειδή βιάζει κατάφορα το δίκαιο το Ισραήλ, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τεθεί τέρμα στην αιματοχυσία των Παλαιστινίων. Εδώ ολοκληρώνονται οι επεξηγήσεις ψήφου για σήμερα. Έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Από το Συμβούλιο έχω λάβει τη θέση του για την πρώτη ανάγνωση μαζί με μια δήλωση επεξηγηματική και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τίτλος θα ανακοινωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης τρίμηνη διορία που διαθέτει το Κοινοβούλιο για να ε, γνωμοδοτήσει αρχίζει αύριο 19 Σεπτεμβρίου 2014. Τα πρακτικά της συνεδρίασής μας θα υποβληθούν προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου και αν δεν έχετε